κυρίσω την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Σήμερα λοιπόν η συνεδρίασή μας θα αφιερωθεί αποκλειστικά σε μια σειρά ψηφοφοριών στο πέρας της οποίας ε, οι συντονιστές ε, θα κάνουν τη δική του συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας αύριο το πρωί στις 9 για δύο ανακοινώσεις μελέτης, μία ε, για τον τρόπο με τον οποίο ε, η συμμετοχή των κρατών μελών μεταφράζεται στον προϋπολογισμό των κρατών μελών και μια δεύτερη ανακοίνωση μελέτης ε, για το πώς λαμβάνεται υπόψη στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισότητα των φύλων. Και μετά έχουμε και μια ανακοίνωση για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης και μετά θα ψηφίσουμε το ψήφισμα σε σχέση με τον προπολογισμό του 2016. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ότι θα γίνει μια έκτακτη ε, συνεδρίαση Budget Lib για τις συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης στις 19 Οκτωβρίου στις 18 και 45 μέχρι τις 20 και 30 αμέσως μετά τον τριμερή διάλογο διότι θα κάνουμε ένα πρώτο ε, τριμερή διάλογο προς συνδιαλλαγής ε, στις 19 Οκτωβρίου αρχές του απογεύματος. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το steering board του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μας ε, κοινοποίησε δύο ονόματα ένα πρώτο που θα οριστεί ως Managing Director, Γενικός Διευθυντής ε, του Ταμείου και ένα δεύτερο όνομα για τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Ταμείου η ακρόση που έχει προβλεφθεί που θα ακολουθηθεί από ε, ψήφο στην Ολομέλεια θα λάβει χώρα αύριο στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάν 6Q2 αύριο στις 7 το βράδυ η συνεδρίαση αυτή μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 2,5 ώρες παρακαλώ λοιπόν να ε, ετοιμαστείτε και φροντίστε να είστε διαθέσιμοι για να ακούσετε αυτούς τους δύο υποψηφίους. Μετά από την καθεμία ακρόαση, ε, καθεμία εκ των οποίων μπορεί να διαρκέσει μία ώρα, θα έχουμε μία με σύντομη ενημέρωση και μετά ψηφοφορία. Και βάσει αυτής της ψηφοφορίας το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει στην Ολομέλεια την Τετάρτη το απόγευμα. θα πρέπει να αποφασίσουμε χωρίς καθυστέρηση διότι το θέμα αφορά την σωστή λειτουργία και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Νομίζω ότι σας είπα τη ε, βασικά σημεία των ανακοινωσεών μου. Περνάμε τώρα λοιπόν στις ψηφοφορίες. Ε, πρώτα απ' όλα για την κινητοποίηση του Μέσο ευελιξίας, την έκθεση της κυρίας Κάτια Ζαμπάλ που έχει σήμερα το απόγευμα δύο εκθέσεις. Να χαιρετήσω την ετοιμότητα και την ε, σαφήνεια ε, με την οποία υιοθετήθηκαν όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ολομέλεια που θα γίνει Τετάρτη απόγευμα. Ε, το διάστημα που θα έχει περάσει θα είναι δύο εβδομάδες, ε, διάστημα ρεκόρ. Και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, την οποία δίνω και το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ακριβώς ε, και σε συνέχεια των όσων είπατε και εσείς για το πόσο γρήγορα διεκπαιρεώθηκαν δύο αυτές εκθέσεις, ήθελα να σας εξηγήσω γιατί στις λίστες ψηφοφοριών εγώ προτείνω ως εισηγήτρια να καταψηφίσουμε όλες τις κατατεθήσεις τροπολές. Ακριβώς γι' αυτό, διότι θεώρησα ότι η ταχύτητα ε, έγκρισης της έκθεσης, δηλαδή πιο ε, ταχεία δυνατή έγκριση της έκθεσης για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση ε, και με τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται είναι υπέρτερο οποιασδήποτε άλλης ιδέας, τροπολογίας. Στο κείμενο εγώ προσπάθησα με τη διατύπωση να μην υπησέλθω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες, αλλά να προσπαθήσω να εκφράσω την άποψη των περισσότερων για να μπορέσουμε, όπως είπα, να εγκρίνουμε τα κείμενα χωρίς τροποποίησης για να τηρήσουμε τις προθεσμίες και να προλάβουμε την Ολομέλεια της Τετάρτης. Αλλιώς δεν θα την προλάβουμε. Υπάρχει και άλλη Ολομέλεια σε 15 ημέρες βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά κατεπήγον ώστε να γίνει αυτή η εξαίρεση και να ψηφίσουμε τις δύο αυτές εκθέσεις χωρίς τροπολογίες να ευχαριστήσω βέβαια τις πολιτικές ομάδες που κατέστησαν τροπολογίες και να τους εξηγήσω ότι δεν είναι λόγο το ότι διαφωνώ επί της ουσίας τι τροπολογίες αυτές, απλά ε, είναι θέμα ταχύτητας, ταχύτερης διεκπαιρέωσης. Γι' αυτό μπήκαν και οι ψηφοφορίες ε, σήμερα στην ημερήσια διάταξη, ώστε την Τετάρτη να μπορέσουν να ψήφουν στην Ολομέλεια. Τι. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, φαντάζομαι ότι αντιλαμβανόμεθα όλοι το κατεπήγον 3 με 5.000 ε, λαθρομετανάστες εξωτερικά σύνορα της Ένωσης κάθε μέρα. Είναι κατεπήγον και πρέπει να κινητοποιηθεί το μέσο και θέλουμε να ε, περιορίσουμε όσο το δυνατόν ε, τις παράνομες εισρωές στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία να βεβαιωθείτε όλοι ότι έχετε βάλει τις κάρτες στα μηχανήματα γιατί μπορεί να χρειαστεί να ψηφίσουμε ονομαστικά ο κύριος Τάραντ. Ε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ε, εγώ ξέχασα την κάρτα μου στο Στρασβούργο, δυστυχώς. Ζητώ συγγνώμη. Ω ένθρωπο υποστηρικτή τη μία έδρα, λέει ο μιλητή. Προτείνει λοιπόν ο πρόεδρο ε, δύο κάρτε να υπάρχουν, μία για το Στρασβούργο και μία για τι Βρυξέλλε. Ώστε να μην ρηψινδυνεύσουμε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, θα ε, έχω το νου μου να κοιτάω την ψήφο σα, κύριε Τεράν, και να την προσθέτω. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντε. Όχι, λείπουν λοιπόν, μερικοί. Εγώ δεν έχω ψηφίσει, λέει ο πρόεδρο. Α, μάλιστα. Πέρα ψηφοφορία, η διάταξη γίνεται δεκτή με τρεις αποχές ο κύριος Ταράν δεν ξέρουμε τι ψήφισε πολύ ωραία λοιπόν έχουμε μια πρώτη τροπολογία παραγραφός 1 τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές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 για το σύνολο τώρα του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ μία κατά δεν υπάρχουν αποχές 24 ψήφους υπέρ συγγνώμη μία κατά Περνάμε στην δεύτερη έκθεση της κυρίας Γκαρδία Ζαμπάλ που, προκύπτει από τις συνέπειες της ψηφοφορίας που μόλις έλαβε ε, χώρα αφορά το σχέδιο διορθωτικού πολυπολογισμού αριθμός 7 που αφορά τις πιστώσεις για την ε, εφαρμογή του ψηφίσματός μας. Των ψηφισμάτων μας περνάμε στην ψηφοφορία ας πάμε τροπολογία 4 υπέρ κατά μπορούμε να ψηφίσουμε σε μπλοκ μαζικά. Όχι. Λοιπόν, υπάρχουν ε, διάφοροι συντάκτες τροπολογιών, οπότε θα ψηφίσουμε μία-μία τις τροπολογίες. Λοιπόν, η 4 απορρίπτεται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές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 3 της ε, G1 νέας ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το σύνολο τώρα του κειμένου του σχεδίου διορθωτικού πολεπολογισμού 7 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ο διορθωτικός προϋπολογισμός εγκρίνεται με 24 ε, ψήφους ε, εναντί και δεν υπάρχουν αποχές. Τώρα λοιπόν πρέπει να προβλέψουμε ορισμένες μεταφορές πιστώσεων. Κυρία Γκαρδιαθάβα, έχετε το λόγο. Δεν έχετε σχόλια. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν σχόλια, Έχουμε μια σειρά, όπως είπα, μεταφορών. Η κυρία Γκαρδιαθάπαλη. Όχι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Η 29 είναι το Global Transfer, το περίφημο, συγκεντρωτική μεταφορά υπολείπου δηλαδή, μετά το τέλος ε, του δημοσιακού έτους. 32 έχει να κάνει με πληρωμές σε σχέση με την ανθρωπιστική κρίση και τους πρόσφυγες για κινητοποίηση του αποθεματικού για επίγουσα βοήθεια 175 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Πρόεδρος, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τις πιστώσεις αυτές ομού, δηλαδή την 29 και την 32, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται λοιπόν 25 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Για τα λοιπά τμήματα. Κυρία Χολμάιερ, δεν έχουν μεγάλη σημασία αυτές τις τροποποιήσεις. Ε, είναι ίσονος ε, επίπτωσης. Ε, θέλετε να μας κάνετε κάποια σχόλια. Λοιπόν, μας έχουν σταλεί οι ε, αποφάσεις των άλλων θεσμικών οργάνων, μόνο για να σας ενημερώσω, να σας πω ότι πρέπει να αποφασίσουμε για το 25, Η τιμή είναι κάτω από τα όρια. Μετά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας έχει υποβάλει τέσσερα ερωτήματα. Το ένα από αυτά αφορά μια μεταφορά κόστους σχετικά με τα παιδιά του προσωπικού που πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Το... Οι μεταφορές αυτές είναι για να καλύψει λοιπόν το κόστος το οποίο έχει αυξηθεί. Το υπαριθμό 102 κεφάλαιο έχει να κάνει με προσωρινή χρηματοδότηση των υπαλλήλων αφότου σταματήσουν να έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου. Είναι κάποιες μεταβατικές πληρωμές 142.000 ευρώ είναι μικρό το ποσό. Έπειτα, μεταφορά υπαριθμών 3 αφορά την αντικατάσταση μηχανημάτων έτσι ώστε να καλύψει λοιπόν διάφορα παροχημένα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εργαστήρια παραγωγής. Υπάρχει ένα ποσό 50.000 ευρώ επίσης για τις ε, εκδόσεις. Αυτές οι γενικές εκδόσεις ανέρχονται σε κόστος 350.000 ευρώ. Είναι μικρό λοιπόν το κόστος. Έπειτα έτοιμα 4 Πρόκειται για ένα ποσό 746.000 ευρώ για τον καθαρισμό και την συντήρηση κτηρίων. Ο στόχος είναι η αντικατάσταση του παροχημένου εξοπλισμού δικτύωσης των εκτηρίων και γενικότερη συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού στον ε, τομέα της πληροφορικής ε, των εκτηρίων. Επόμενο αίτημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, αυτό αφορά και κάποιες προσωρινές ενισχύσεις των ευρωβουλευτών. Η πρόταση που υπέβαλε το Δικαστήριο είναι εξαιτία της αύξηση του φόρτου εργασία να αυξηθούν και οι γλωσσομαθείς νομικοί, οι οποίοι θα αναλάβουν μεταφράσεις. Η αιτιολόγηση λοιπόν από το δικαστήριο είναι αυξημένος φόρτος εργασίας και ανάγκη αύξησης του αριθμού των ε, εσωτερικών και εξωτερικών ε, μεταφραστών. Αυτά λοιπόν ε, προς το παρόν είναι ενημερωτικά τα περισσότερα αυτά που έχω να σας πω. Εκτός μικροφώνου Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σιωπηρά εγκρίνονται. Αν δεν έχετε αντίρρηση με βάση το άρθρο 25 του κανονισμού. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στην Επιτροπή των Περιφερειών. Επίσης ε, εδώ υπάρχει μια περίπτωση του άρθρου 25. Χρειάζονται λίγο λιγότερα χρήματα εδώ για τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, για τις πολιτικές τους ε, δραστηριότητες, όμως χρειάζεται αύξηση των κονδυλίων έτσι ώστε να συσταθεί ένα αυτόματο σύστημα μετάφρασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά των ε, πληροφοριών από εδώ εκεί, έτσι όπως λέει το κείμενο στα αγγλικά, για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αυτόματης ε, μετάφρασης ε, πολλαπλών πηγών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των μεταφραστικών εργασιών. 200.000 λοιπόν, είναι λίγο πάνω από το όριο. Έπειτα, τρίτον, υπάρχει το ελεκτικό συνέδριο. Το οποίο υπό τις γενικότερες διατάξεις ζητεί πρόσθετα κονδύλια για υπηρεσίες μετάφρασης έχουν αυξηθεί ανάγκες του σε μετάφραση. Η αιτιολόγηση είναι παρόμοια με εκείνη του δικαστηρίου, ότι δηλαδή η μείωση του προσωπικού έχει οδηγήσει σε ανάγκη ε, πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών. Μετά, μετατροπή και αντικατάσταση των ε, εστιατορίων. Πρέπει να γίνουν κάποιες ε, εργασίες ανακαίνιση στην καφετέρια, στα έπιπλα, 40.000 ευρώ εδώ. Χρειάζονται διάφορα ε, εργασίες αντικατάστασης, εργονομικά τραπέζια, κάτι το οποίο έχει ζητηθεί κατόπιν σύστασης ιατρών. Έπειτα, αγορά νέου εξοπλισμού και εγκατάσταση αυτού 65.000 ευρώ για πρόσθετο εξοπλισμό. έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των εργασιών του ελεκτικού συνεδρίου. Συνολικό ποσό 220.000 ευρώ, το οποίο θα αφαιρεθεί από τους βασικούς μισθούς. Αυτά. Merci, Σας ευχαριστούμε, κύριε Συγγήτρια. Πέντε λοιπόν αιτήσει μεταφοράς ε, ε, έχουμε για το δικαστήριο, μία για την Επιτροπή των Περιφερειών ε, και μία αίτηση από το Ελληνικό Συνέδριο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε, εκτός αν το επιθυμεί κάποιος από εσάς, γιατί το Αφρικό 25 του κανονισμός επιτρέπει εάν δεν τεθούν σε ψηφοφορία, να θεωρηθούν σιωπηρός εγκεκριμένε οι αιτήσει. Δεν βλέπω κάποια αντίρρηση, επομένως θεωρούμε ότι αυτές οι αιτήσει μεταφοράς ε, που μας εκτέθησαν υπόψη γίνονται ομόφωνα δεκτές από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όσον αφορά την κεντριακή πολιτική δεν υπάρχουν αιτήματα και έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Υπό τα διάφορα υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο τον λόγο. Τερματίστε τη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί στι 9. Και καλό του συντονιστέ να παραμένουν. Θα συνεχίσουμε τι εργασίε μα σε 5 λεπτά.